Λοιπόν, αγαπητοί συναδελφοί, καλώς ήρθατε στο τελευταίο κομμάτι τη συνεδρίασής μας πριν τις διακοπές. Έχουμε ένα σημαντικό θέμα στην μερίσια διάταξη, το οποίο είναι η Πολωνική Προεδρία στον τομέα της υγείας και είναι Μεγάλη μου χαρά να καλωσορίζω την κυρία Υπουργό, την κυρία Εύα Κόβατς. Καλώς ήρθατε. Είστε υπεύθυνοι για την πολιτική υγεία στην Πολωνία και ε, πρόεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτών. Είστε καλοδεχόμενοι εδώ πέρα στην Επιτροπή Κλιματικής ε, Προστασίας αλλά και Προστασίας Υγείας. Και εμείς είμαστε υπερήφανοι για το ότι πέρα από το περιβάλλον ασχολούμαστε και με την υγεία. Και νομίζω πως ε, όταν το οργανώναμε τότε μάλλον θα θεωρούσαν πως η ρήπανση είναι και κίνδυνος για την υγεία, γι' αυτό τα κανονίσαν έτσι. Γι' αυτό η Επιτροπή λέγεται Περιβάλλοντος και Υγείας. Ε, εν τω μεταξύ βεβαίως έχει αποκτήσει και άλλες αρμοδιότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολίτες αναμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση διάφορες δραστηριότητες για πρόληψη εναντί κινδύνων της υγείας, για κοινέ πρωτοβουλίες, για τις μεγάλες ε, ασθένειες, για την έρευνα, αλλά και για πρακτικά ζητήματα. για να παραμένουν υγιείς. Έχουμε εδώ πέρα διάφορα νομοθετικά θέματα. Τον αγώνα κατά της ε, πειρατείας ε, φαρμάκων το θέμα της φαρμακοεπαγρύπνησης των παρενεργειών των φαρμάκων, την διασυνοριακή παροχή υγείας και το μεγάλο φαρμακευτικό πακέτο το οποίο θα απασχολήσει και την Προεδρία σας. Πέρα από την Επιτροπή Εξωτερικών, η δική μας είναι η δεύτερη πόλη υπάρχει και μια ομάδα εργασίας για την υγεία. Οι συνάδελφοι που είχαν εργαστεί δηλαδή σε αυτόν τον τομέα και πλέον είναι έμπειροι και συμμετέχουν εδώ μέσα. Και εσείς έχετε σπουδάσει βλέπω ιατρική, είστε του κλάδου και χαιρόμαστε. Πού σας ε, βλέπουμε εδώ πέρα. Ε, ελπίζουμε να μας εξηγήσετε το πρόγραμμα της ε, Πολωνικής Προεδρίας. Καλώς ήρθατε και έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που μου δίνεται ευκαιρία να σταθώ μπροστά σας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας στα θέματα της υγείας. Δεν κρύβω την είναι ιδιαίτερη στιγμή. Αφενός λόγω του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ενισχύθηκε σημαντικά μετά τη θέση ισχύ της Σύνθηκης της Λισαβόνας και αφετέρου λόγω της προσωπικής σας προσήλωσης σε σημαντικά και οικία για τον πολίτη θέματα όπως είναι τα θέματα που αφορούν την υγεία. Με την έναρξη της Πολωνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινά ταυτόχρονα και η εφαρμογή του νέου προγράμματος 3, στα πλαίσια του οποίου η Πολωνία θα έχει τη χαρά να συνεργαστεί με τη Δανία και την Κύπρο. Οι εργασίες μας θα στοχεύσουν τόσο στην βελτίωση της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών, όσο και στην προστασία των ευρωπαϊκών κοινωνιών από κοινού παράγοντες κινδύνου. Επιπλέον, στο σχέδιό μας, πρώτα απ' όλα θα επικεντρωθούμε στην εξασφάλιση ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης για τους Ευρωπαίους πολίτες. Τρία είναι τα κύρια θέματα του προγράμματος ε, τρίο, των τριών προεδριών για τα θέματα υγείας. Πρώτον, η μη λιμώδης νόση και η υγιής γύρανση. Δεύτερον, οι ασθένειες χωρίς σύνορα και άρα και η υγειονομική ασφάλεια. Και τρίτον, καινοτομία και καλές πρακτικές. Τα θέματα αυτά δεν συνεχίζουν μόνο τις εργασίες των προηγούμενων προεδριών, αλλά συνδέονται και με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2006 για τις κοινέ τιμές ε, για κοινέ αξίες και αρχές ε, της ε, υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα εντάσσονται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία και στη στρατηγική Ευρώπη 2020. Κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, οι προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας για την υγεία αποτελούν τμήμα του προγράμματος ε, των τριών προεδριών, του τρίου. Δύο είναι οι βασικές προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας για την υγεία που σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε. Πρώτον, η μείωση των διαφορών στην υγεία μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και η πρόληψη εγκεφαλικών παθήσεων και νευροεκφυλιστικών παθήσεων όπως την όσο του Αλσχάιμερ. Στα πλαίσια της πρώτης προτεραιότητάς μας Πρώτα απ' όλα θα τονίσουμε την ανάγκη μείωση των διαφορών στην υγεία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ό,τι αφορά τους καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία. Παρόλο που οι υπηρεσίε υγείας είναι προσιτές σε όλους τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημαντικές και αποδεδειγμένες ανισότητες στην υγεία μεταξύ των χωρών μελών. Αυτές οι διαφορές εντοπίζονται ακόμη και στο εσωτερικό της ίδια χώρα. Σήμερα 80% του συνόλου των θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλεται σε χρόνιες μη λοιμώδεις νόσους. Αυτές ε, επιβαρύνουν όλο και περισσότερο τις δαπάνες υγείας των διαφόρων χωρών μελών. Η λοιμώδης νόση ήταν άλλοτε η κύρια αιτία θανάτου. Σήμερα όμως τελούν υπό έλεγχο και προκαλούν λιγότερο από το 2% των πρόωρων θανάτων. Η εμφάνιση χρόνιων μη λιμοδονώσεων, όπως ε, οι παθήσεις του κυκλοφοριακού ή του αναπνευστικού συστήματος, πολλοί καρκίνοι και διαταραχές του μεταβολισμού, όπως ο διαβήτης, συνδέονται όλο και περισσότερο με τέτοιους παράγοντες κινδύνου, όπως είναι το κάπνισμα, η ακατάλληλη διατροφή, η έλλειψη σωματικής άσκησης και η κατάχρηση νοπνεύματος. Η καταπολέμηση των διαφορών στην υγεία αποτελεί σημαντική πρόκληση. Βέβαια, οι σημερινές δράσεις και τα μέτρα που θα λάβουμε θα αποφέρουν καρπούς μακροπρόθεσμα μόνο. Παρόλο που γνωρίζουμε τις αρνητικές συνέπειες του καπνίσματος και της καθιστικής ζωής, είναι δύσκολο να αλλάξουμε τις κακές μας συνήθειες ή τον τρόπο ζωής μας. Το κάπνισμα είναι η κυριότερη αιτία πρόωρων θανάτων που μπορούμε κάλλιστα να αποφύγουμε. Η νοικοτήνη προκαλεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θάνατο περίπου 650.000 πολιτών ετησίως. Το 25% δηλαδή του συνόλου των πρόωρων θανάτων. Άλλος παράγοντας με τεράστια σημασία για την υγεία των Ευρωπαίων είναι το ινόπνευμα. Πάνω από το 13% των πρόωρων θανάτων ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλεται σε κατάχρηση ινοπνεύματος. Η κατάχρηση ινοπνεύματος συνεπιφέρει και κοινωνικά αποτελέσματα εκτός από τα προβλήματα στην υγεία που επιβαρύνουν το σύνολο της κοινωνίας ε, εκτός από τις μεμονωμένες οικογένειες. Θεωρούμε επιτακτική ανάγκη τη σύσφυξη της συνεργασίας ε, για τα θέματα αυτά μεταξύ των κρατών μελών. Άλλο πρόβλημα δημόσιας υγείας που θα προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε ως σημαντική προτεραιότητα της Πολωνικής Προεδρίας είναι η έξαρση του φαινομένου της παχυσαρκίας και του υπερβολικού βάρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το φαινόμενο αυτό έχει λάβει πια τις διαστάσεις επιδημίας, με ιδιαίτερα ανησυχητική την εμφάνισή του σε παιδιά και νέους. Το ποσοστό των παχύσαρκων στον κόσμο διπλασιάστηκε τα τελευταία 30 χρόνια. Το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία αποτελούν την πέμπτη αιτία θανάτων και αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγκιακών παθήσεων, παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος, καρκίνων, διαταραχές του μεταβολισμού, όπως διαβήτη κτλ. Πρόσφατα στοιχεία μας δείχνουν ότι από υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία υποφέρει το 17 ε, εκατομμύρια νέων Ευρωπαίων. Έχουμε υπόψη ότι η παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος δεν είναι μόνο ε, ιατρικό πρόβλημα, αλλά δημιουργεί και τεράστιες οικονομικές προκλήσεις, γιατί προκαλεί κατακόρυφη αύξηση των δαπανών της ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οι καθοριστικοί παράγοντε της υγείας που οδηγούν στις ανισότητες μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών αποτελούν σημαντική πρόκληση της δημόσιας υγείας. Γι' αυτό και επιλέξαμε αυτό το θέμα ως μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας. Θέλουμε επίσης ε, να επισημάνουμε την ανάγκη πρόληψης, έγκαιρης αντιμετώπισης, διάγνωσης και ελέγχου των νόσων του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά. Οι χρόνιες μη λιμώδεις ε, παθήσεις του αναπνευστικού είναι από τις πιο συχνές ασθένειες της παιδικής ηλικίας και η συχνότητα εμφάνισής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη, ανέρχεται κατά μέσο όρο από 10-30% επαθείς αυτές ε, επηρεάζουν αισθητά την ποιότητα ζωής. Επιδεινώνουν τη φυσική κατάσταση και την ικανότητα συγκέντρωσης, επιδρούν αρνητικά στην ανάπτυξη του παιδιού και πολύ συχνά οδηγούν και στην κοινωνική του περιθωριοποίηση. Η βλάβη των αναπνευστικών οδών στη διάρκεια της παιδικής ηλικίας αυξάνει και το κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων πνευμονοπαθήσεων και, και καρδιοπαθειών. Ε, αυτές οι χρόνιες ε, ασθένειες μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε αναπηρία ή πρόωρο θάνατο. Η έγκαιρη διάγνωση, η πρόληψη και η παρακολούθηση των μη λιμωδών νόσων του αναπνευστικού, ιδιαίτερα σε νέους και παιδιά, μπορούν να περιορίσουν τις αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές ε, συνέπειες που συνδέονται με τις νόσους αυτές και να επιδράσουν θετικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Κυρίες και κύριοι, στη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας θα θίξουμε και το ζήτημα της έγκυρης διάγνωσης και θεραπείας των επικοινωνιακών διαταραχών στα παιδιά και την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής υγείας και κάποιων νεοτεριστικών καινοτόμων λύσεων. Γνωρίζουμε ότι η σωστή λειτουργία των οργάνων ακοής, όρασης και ομιλίας αποτελεί τη βάση της, οικονομ... της κοινωνικής επικοινωνίας και της ανάπτυξης της σύγχρονης κοινωνίας της πληροφορίας. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναλάβουμε δράσεις που θα επιτρέψουν την έγκαιρη διάγνωση των δυσλειτουργιών ε, των αισθητηρίων οργάνων και να εφαρμόσουμε έγκαιρα θεραπεία και αποκατάσταση. Σε πολλές χώρες μέλη, εδώ και μερικά χρόνια, γίνονται διάφορες προσπάθειες με στόχο τη διάδοση του προσυμπτωματικού ελέγχου του, της ακοής, όρασης και ομιλίας στα παιδιά με έγκαιρη διάγνωση των επικοινωνιακών διαταραχών και κατάλληλη ιατρική παρέμβαση, καθώς και με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής ε, υγείας και των όβων τεχνολογιών, μπορούμε να εξασφαλίσουμε σωστή ανάπτυξη στα παιδιά. Και αυτό θα έχει τεράστια επιρροή στην ποιότητα ζωής τους και στο μέλλον μπορεί να βελτιώσει την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική τους κατάσταση. Έχουμε επίσης ε, επίγνωση των ε, προσπαθειών που έγιναν στον τομέα αυτό στο Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής υγείας. Στα πλαίσια αυτών των τριών ε, θεμάτων, προκειμένου να μειώσουμε τις ανισότητες στην υγεία των Ευρωπαίων πολιτών, θεωρούμε αναγκαία την εφαρμογή προγραμμάτων προς συμπτωματικού ελέγχου και την ανάγκη δημιουργίας δικτύων μεταξύ των διαφόρων Ιδρυμάτων Υγείας για την παρακολούθηση των φαινομένων της υγείας. Θα επικεντρωθούμε στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, ιδιαίτερα στην ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών. Πιστεύουμε ότι η έγκαιρη αντιμετώπιση από την παιδική ηλικία μιας αρρώστιας εξασφαλίζει πολύ καλύτερη ζωή στο μέλλον και μάλιστα βοηθάει για την καλύτερη εξασφάλιση των ίσων ευκαιριών. Ας μην ξεχνάμε ότι η υγιής γύραση αρχίζει με την υγιή παιδική ηλικία. Για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων μας πρόκειται να οργανώσουμε και μία σειρά διασκέψεων εμπειρογνωμόνων και μία υπουργική διάσκεψη με τον τίτλο η μείωση των διαφορών υγείας στις χώρες μέλη. Θα λάβει χώρα η υπουργική αυτή διάσκεψη στο Πόσναν της Πολωνίας 7 και 8 Νοεμβρίου του 2011. Στα πλαίσια των προτεραιοτήτων μας για τις παθήσεις των ηλικιωμένων θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες προκειμένου να προλάβουμε να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα και να θεραπεύσουμε εγκεφαλοπάθειες ή νευροεκφυλιστικές παθήσεις όπως την όσο του Αλτσχάιμερ. Στη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας δώσαμε έμφαση στην υλοποίηση και στήριξη εθνικών πολιτικών υγείας. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να προσδιορίσουμε τις οργανωτικές και οικονομικές ανάγκες και τις προκλήσεις ε, όπως, την, ε, τον, όπως ο αυξανόμενος αριθμός ε, ηλικιωμένων και ο αυξανόμενος αριθμός παθήσεων ηλικιωμένων από αρρώσκες που είναι χαρακτηριστικές για την προχωρημένη ηλικία, όπως είναι η άνοια ή οι νευροεκφυλιστικές ε, παθήσεις. Θα αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία στη μελέτη του εγκεφάλου σε καινοτόμες ε, διαγνωστικές μεθόδους, στη θεραπεία και στην παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας στους ηλικιωμένους που νοσούν από τέτοιες ασθένειες, ενώ θα επικεντρωθούμε και στην αφύπνιση του κοινού για θέματα υγείας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η προτεραιότητα αυτή ακολουθεί και προηγούμενες προσπάθειες και ενέργειες Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εταιρική σχέση στην καινοτομία στα πλαίσια της υγιούς και ενεργούς γύρανσης. Η υλοποίηση, για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων μας αυτών θα οργανώσουμε και μια διάσκεψη εμπειρογνωμόνων με τον τίτλο «Η πρώτη Ευρωπαϊκή ημέρα του εγκεφάλου. Γύρανση, εγκεφαλικό επεισόδιο και νόσος Ολχάιμερ. Αναζήτηση καινοτόμων λύσεων. διάσκεψη αυτή θα λάβει χώρα στην Βαρσοβία στις 18 Νοεμβρίου του 2011. Στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Σόποτ, ξεκινήσαμε τον πολιτικό διάλογο με τους Υπουργούς Υγείας. Πριν από δύο μέρες ξεκίνησε τις εργασίες της και η ομάδα εργασίας για θέματα δημόσιας υγείας, στην οποία υπευλήθη ένα σχέδιο συμπερασμάτων για την πρόληψη και θεραπεία των ε, επικοινωνιακών διαταραχών στα παιδιά, ενώ υπευλήθηκε το πρόγραμμα εργασιών της Πολωνικής Προεδρίας. Η Πολωνική Προεδρία προτίθεται να προτείνει στο Συμβούλιο Υπουργών και συμπεράσματα με θέμα την εξάλληψη των διαφορών στην υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω κάποιων δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τους καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία και προσπάθεια έγκαιρης αντιμετώπισης και ελέγχου μη λιμωδών νόσων του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να τονίσω και να διατρανώσω ότι είμαστε ανοιχτοί και πρόθυμοι να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτηση και να συζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα σας ενδιαφέρει. Προσβλέπουμε σε καρποφόρα συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα πλαίσια των εργασιών επί των νομοθετικών πρωτοβουλειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στα πλαίσια του τριό, ήδη ε, στην αρχή της Προεδρίας απέθυνε, έκκληση στον πρόεδρο Νταλή ε, για να εγκριθεί ένας οδικός χάρτης ε, με τις προτεραιότητες που θα υλοποιήσουμε. Επιλέγοντας τις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας θέλουμε να δείξουμε ότι η υγιής παιδική ηλικία είναι το πρώτο βήμα για μια υγιή και δραστήρια τρίτη ηλικία. Έχω την ελπίδα ότι οι προτάσει μα θα γίνουν δεκτέ και από εσά, αλλά θα τι αναγνωρίσει και η ευρωπαϊκή κοινωνία. Άλλωστε, εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη βελτίωση της κατάστασης υγείας στην Ευρώπη. Η αλληλεγγύη είναι για μας πολύ σημαντική και όχι μόνο από ιστορική άποψη. Σημαντική είναι και μια άλλη διάσταση της αλληλεγγύης. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην υγεία. Και τέτοια αλληλεγγύη θέλουμε να αναπτύξουμε στην Ευρώπη. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την προσοχή σας και να σας είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Äh, Κυρία Υπουργέ, ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση των βασικών σημείων της ε, Πολωνικής Προεδρίας. Ενδιαφέροντα πράγματα αυτά τα οποία μας είπατε. Πράγματι, το πρόγραμμα μέτρων για την υγεία, στην παιδική ηλικία, έχετε δίκιο, αν μεγαλώσουν υγιεί τα παιδιά είναι μεγάλη πιθανότητα να παραμείνουν και υγιεί. Έχουν μπει σωστές ρίζες δηλαδή. Μετά αναφέρατε τα προληπτικά μέτρα τα οποία μπορούμε να λάβουμε σε εξαρτήσεις όπως ε, το ενόπνευμα, ο καπνός, ε, όπου αναμένουμε μια νέα οδηγία της Κομισιόν και βεβαίως το ότι καθόμαστε και τρώμε όλη μέρα και αυτός ο τρόπος ζωής ε, πρέπει να αλλάξει και να κινηθούμε λίγο περισσότερα γιατί αυτός είναι ο φθηνότερος τρόπος να εξοικονομήσουμε λεφτά και να μην αρρωσταίνουμε. Μετά αναφέρατε αρκετά θέματα που είναι και για μας σημαντικά, ειδικά όσον αφορά τις ε, ασθένειες των ηλικιωμένων. Γινόμαστε πιο ηλικιωμένοι γενικά στην Ευρώπη και είναι θέμα που μας αφορά. Είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον πως μόνο 2% των ασθενειών είναι μεταδοτικές. Πριν 100 χρόνια ήταν διαφορετική η κατάσταση. Σήμερα είναι άλλες οι ασθένειες, διαβήτης, καρκίνος. Όλες αυτές οι αρρώστιες του δυτικού πολιτισμού που ξέρουμε. Οι συνάδελφοι έχουν τώρα αρκετές ερωτήσεις. Ξεκινάμε με τον κατάλογο των ομιλητών. Πέτερ Λίζε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου. Ε, εγώ έχω απογοητευτεί λίγο λόγω του, της ώρας, γιατί δεν είμαστε τόσο πολλοί, αλλά σας πω πως οι συνάδελφοι ε, της πολωνικής πλατφόρμας, βλέπετε πέρα, εκπροσωπούνται ε, με έξι άτομα. Οπότε οι υπόλοιποι συνάδελφοι μπορεί να μην έχουν έρθει, αλλά από την πολωνική πλατφόρμα είναι εδώ πέρα. Διάβασαμε ενδιαφέρον πώς και εσείς, όπως και εγώ, είχατε ασχοληθεί με την παιδιατρική. Ξέρετε πως έχουμε επίσης μια ομάδα διακομματική στο Κοινοβούλιο για τα πρόωρα νεογνά για να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερη φροντίδα. Εμείς μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό το θέμα κάποια στιγμή. Ε, κάποιες ερωτήσεις τώρα. Πρώτα απ' όλα, το είπε και ο πρόεδρος, φαρμακευτικό πακέτο δεν έχει κλείσει. Αναμένουμε τις ερχόμενες εβδομάδε την αλλαγμένη πρόταση της Κομισιόν για την πληροφόρηση των ασθενών. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να υποστηρίξετε αυτά τα οποία θέλει το Κοινοβούλιο στο Συμβούλιο. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να είναι πιο ευανάγνωστο το χαρτί που συνοδεύει τα φάρμακα και δεύτερον να υπάρχει ένα κουτάκι που με λίγα λόγια θα περιγράφει το φάρμακο. Γιατί οι περισσότεροι ασθενείς δεν διαβάζουν όλο αυτό το χαρτάκι και δεν ξέρω αν θέλουμε να το διαβάσουν. Γιατί ε, πανικό θα πάθουν μόνο εάν το διαβάσουν όλο. 5-6 σημεία βασικά. Και ανεξαρτήτως ε, των πληροφοριών από την φάρμακοβιομηχανία μπορούν να υπάρξουν βάσεις δεδομένων από τρίτους, είτε τις εθνικές αρχές, είτε κάποιους άλλους που δεν είναι φαρμακοβιομηχανίες για να ενημερώνουν ανεξάρτητα. Δεύτερο θέμα ε, τους ε, δωρητές ε, γιατί είχαμε μια πρωτοβουλία χτες για τους ε, εθελοντές δωρητές βεβαίως, οι οποίοι δεν θα αμείβονται. Είχαμε νομίζω αρκετά καλά αποτελέσματα για τους δωρητές οργάνων και στη Λισαβόνα αναφέρεται πως ε, δεν επιτρέπεται να αποτελέσει αντικείμενο εμπόριο μέρος του ανθρωπίνου σώματος, αντικείμενο εμπορίου. Και δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί κάτι σχετικά για να το φέρετε το θέμα αυτό στο Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ, Λίντα Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Υπουργέ που ήρθατε εδώ σήμερα. Τονίσατε ορισμένα πάρα πολύ σημαντικά θέματα για την ευρωπαϊκή υγεία. Άκουσα είπατε για τις ελληνικές ε, νόσους. Υπάρχει μια πολύ σημαντική διάσκεψη στις ΗΠΑ και θα βάλουμε στη δική μας ατζέντα το Σεπτέμβριο ε, μια ημερομηνία για την προετοιμασία αυτή της διάσκεψης του ΕΕ. Άκουσα και τι είπατε για τις ε, νοητικές διαταραχές. Ε, πρόσφατα αρχίσαμε να κάνουμε έρευνα για αυτές τις νοητικές διαταραχές, για τις εγκεφαλοπάθειες. Το θέμα είναι ποια είναι η προσθεμένη αξία του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αυτά. Έτσι λοιπόν έχουν περάσει πολλές προεδρίες από εδώ, ε, αναφέρονται διάφορα ζητήματα, αλλά έρχονται πολίτες και μου λένε και τελικά ποιο είναι το αποτέλεσμα ε, και οι πολίτες απογοητεύονται γιατί δεν υπάρχει κοινό σκεπτικό. Λέμε περίμετως χάρη, καθοριστικοί παραγοντές για την υγεία είναι ζωτική σημασία, όμως δυστυχώς ε, υπάρχουν κάποια θέματα επί των οποίων δεν μπορούμε να εμπνευσούμε τα θέματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παραδείγματος χάρη στο Συμβούλιο Συμβουλίου των Υπουργών δεν βρίσκουμε υποστήριξη για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα έτσι όπως πρέπει. Δηλαδή έχουμε άσκηση πίεσης ε, από ε, τη βιομηχανία, από το κλάδο και δεν είμαστε τόσο αυστηροί όσο θα έπρεπε. Δηλαδή μιλάμε για τα θέματα αυτά για την υγεία αλλά δεν καθορίζουμε από, κοινά, από κοινού τις πολιτικές ε, συζητήσαμε και το θέμα της ε, κοινή αγροτικής πολιτικής και της κοινή ελευθερικής πολιτικής. Θα υπάρχει αναθεώρηση των δύο αυτών πολιτικών σε επόμενους μήνες. Εγώ Με λοιπόν ε, πώς ε, βλέπετε τη δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βάλει ως προτεραιότητα τα θέματα για την υγεία. Αντωνία Παβανόβα. Αντωνία Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Υπουργέ. Εδώ είμαι. Εκτιμώ το φιλόδοξο πρόγραμμά σας. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, να μην επαναλάβω αυτά τα οποία ρώτησαν οι συνάδελφοι. Αναφέρατε τη μείωση του κενού της ανισότητας της υγειονομικής των Ευρωπαίων πολιτών. Είχαμε και μία ακρόαση και βεβαίως σε έξι μήνες δεν μπορείτε να λύσετε προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί εδώ και γενιές, δεκαετίες. Τότε οι ανισότητες επηρεάζονται και από οικονομικές και οικονομικές κρίσεις. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σκοπεύετε να κάνετε μια συζήτηση για την οικονομική βιωσιμότητα των στήματων υγείας. Γιατί τα δεδομένα δείχνουν πως όλα ανεξαιρέτως τα κράτη-μέλη ε, πρώτα απ' όλα άρχισαν να κόβουν από την υγεία. Και από όσο ξέρουμε, ο Επίτροπος Υγείας, ε, ως πρώην Υπουργός Υγείας ε, και Οικονομικών, σκοπεύει να ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση και να δει πώς θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε την βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας Σκοπεύετε λοιπόν να ξεκινήσετε κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ. Ε, υπάρχει ηχό εδώ μέσα. Δεν ξέρω αν είναι τεχνικό το πρόβλημα, αλλά ακούγεται ωραία. Yeah, ακούω, ακούω τη φωνή σας διπλή, δεν ξέρω αν... Και δεν έχω πιει κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, Κάλεμπαχ. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ ε, για το ότι θέσατε τις παιδικές ασθένειες στις προτεραιότητές σας. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, αυτή τη στιγμή έχουμε την ευτυχή κατάσταση στην Ευρώπη, ότι μόνο 2% των θανάτων οφείλεται σε μεταδοτικές ασθονίες. Αυτό δεν είναι τυχαίο όμως, δεν είπα ότι έχουν εξαλειφθεί αυτές οι ασθένειες, απλά τα τελευταία χρόνια ή πριν από μερικά χρόνια υπήρχε ε, μεγάλο ποσοστό εμβολιασμού και έχει υπάρξει μια αλυσίδα εφοδιασμού και παρόλα αυτά αρέστιες οι οποίες θα έπρεπε να έχουν εξαφανιστεί το 2010 εξακολουθούν να υπάρχουν και να αυξάνονται στην Ευρώπη. Οπότε εγώ φοβήθηκα με αυτό το οποίο είπατε που λέτε πως είναι υποέλεγχο οι μεταδοτικές ασθένειες στην Ευρώπη. Εγώ φοβάμαι που συμβαίνει το αντίθετο και νομίζω πως Υπήρχε και μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσκεψη επί Ουγγρικής Προεδρίας στη Βουδαπέστη που τόνισε αυτό το ζήτημα και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δώσετε βάρος ξανά στον εμβολιασμό, ειδικά στην παιδική ηλικία. Θα ήταν λάθος αν αυτή την επιτυχία δέκα ετιών, επειδή ε, βρισκόμαστε σε μια λανθασμένη εντύπωση πως είμαστε ασφαλείς, να την διακινδυνεύσουμε. Ευχαριστώ. Μπορούς Λαυσόνικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, καταρχήν, ε, σε ό,τι αφορά τα νέα ψυχοφάρμακα, τα designer drugs που κατέκλυσαν τα τελευταία χρόνια τις ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται για ψυχοφάρμακα που πολλώνται νόμιμα σαν αντικείμενα συλλογής και οδηγούν αυτά τα designer drugs, αυτά τα τεχνικά ναρκωτικά σε πρόωρους θανάτους. Και μάλιστα η Πολωνία έθεσε αυτό το ζήτημα με ριζικό τρόπο το ρύθμισε, απαγορεύοντας ε, τη χρήση τέτοιων designer drugs ε, θέλετε να προωθήσετε μια τέτοια πανευρωπαϊκή απαγόρευση για να γενικευθεί η πολωνική ρυθμίση και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, σε ό,τι αφορά την οδηγία για την απαγόρευση του καπνίσματος και την εξάρτηση από την νοικοτήνη, ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα σχέδια είναι η εισαγωγή ενιαίας συσκευασίας για τα πακέτα σιγαρέτων. Βέβαια, κάτι τέτοιο μπορεί να είναι, αντι... να είναι παράνομο, να αντιβαίνει στο δίκαιο. Αυτή την επίθεση ακούσαμε μέχρι στιγμής. Εμείς ε, πιστεύω θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προωθήσουμε ένα τέτοιο μέτρο στο μέλλον. Ο κύριος Κρήτον Αρσένης. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να σας καλωσορίσω, κύριε Υπουργέ, στην ε, Επιτροπή μας. Έχω μια ερώτηση. Χάρηκα πάρα πολύ, ικανοποιήθηκα πολύ που άκουσα την ομιλία σας και είδα και τις δραστηριότητες της Προεδρίας σας, το πρόγραμμά σας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που επικεντρώνεστε στην υγεία του ατόμου και στην ε, διατροφή. Ε, το, η νομοθεσία για τα νέα τρόφιμα, novel food, είναι πάρα πολύ σημαντική για μας εδώ στο Κοινοβούλιο και φέτος ακριβώς ε, είχαμε διαφωνία με το Συμβούλιο γιατί ε, θέλαμε να απαγορεύσουμε τα προϊόντα από κλωνοποιημένα ζώα. Δεν θέλαμε να φτάσουν στο πιάτο μας. Έτσι λοιπόν θέλω να ρωτήσω ποια είναι η δική σας θέση για το θέμα αυτό και αν ε, θα υποστηρίξετε την πρόταση της Κομισιόν. Επίσης, ένα άλλο θέμα που είχαμε στο θέμα της διασυνοριακής υγείας ήταν το θέμα των ε, λουτροθεραπείων, οι οποίες ε, μπορούν να οδηγήσουν στην πρόληψη ε, κάποιων νόσων και επίσης ε, είναι και ζωτική σημασία για την άπτυξη των οικονομιών μας. Ευχαριστώ, Αλουίς Πέτελε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ που παρουσιάσατε τους φιλόδοξους στόχους της Πολωνικής ε, Προεδρίας και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την έμφαση που δώσατε στην πρόληψη ειδικά σε σχέση με τους νέους. Εγώ θεωρώ πως ε, πραγματικά χρειάζεται τέτοια στρατηγική αντιμετώπιση Πρέπει να έχουμε περισσότερους υγιείς ανθρώπους γιατί έτσι θα μειωθεί η ροή των νέων ασθενών. Χαίρομαι για το ότι στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Υγείας, στην έκθεση που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο είπαμε πως χρειαζόμαστε την, υγεία, την υγεία σε όλες τις πολιτικές και υγεία για όλους. Αλλά ξέρουμε πως τα κράτη-μέλη έχουν προβλήματα με τα συστήματα υγείας. Από την άλλη οι πολίτες περιμένουν περισσότερα από το κράτος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ξέρουμε ταυτόχρονα πως τα κράτη δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πολιτών. Να αναφέρω λοιπόν πως μιλήσατε για αλληλεγγύη και θα ήθελα να σας πω τι μου συνέβη εμένα όταν συνάντησα μια ομάδα ανθρώπων που ήθελαν να αναπτύξουν έναν υγιή τρόπο ζωής. Με ρωτήσανε είμαστε υποχρεωμένοι να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σε αυτούς που ζουν διαφορετικά και δεν σέβονται κάποιους κανόνες. Το ερώτημά μου είναι, θεωρείτε πως οι ασφάλειες, η υγείας θα μπορούσαν να προσέχουν περισσότερο αυτό το θέμα. Οι άνθρωποι δηλαδή που ασχολούνται με την υγεία τους ε, να κερδίσουν και κάτι. Όπως συμβαίνει με τους οδηγούς παραδείγματος χάρη. Εάν ε, δεν τρακάρει κανείς για ένα χρόνο μειώνεται το ασφάλιστρο. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο, πώς βλέπετε τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Πολλοί στόχοι, νομίζω, θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω της στήριξης της κοινωνίας των πολιτών. Αντί για... από το Υπουργείο Υγείας. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία για αυτό το εξάμεινο. Ευχαριστώ. Πολύ λεπτή ερώτηση. Όταν είσαι άρρωστος σε τιμωρεί και η ασφάλεια. Και όταν δεν είσαι άρρωστος παίρνεις πόντους. <laughs> Ε, θα απαντήσει η κυρία Υπουργός. Εντίτε στρέλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Υπουργέ. Και εγώ θα ήθελα ε, να αναφερθώ σε αυτά τα πολύ σημαντικά στο οποίο αναφέρατε, στον μυθισμό, στο αλκοόλ και στο κάπνισμα, σε ζητήματα που σχετίζονται με την παχυσαρκία και αναφερθήκατε στην αναγκαιότητα να διασφαλίσουμε έναν υγιή τρόπο ζωής για τα παιδιά εξαπαλώνων ήχων. Εγώ ήμουν εισηγήτρια στην Επιτροπή αυτή για την έκθεση για τις ανισότητες στην υγεία. Και κατά την ε, ανάλυση που έκανα και στην πρόταση που παρουσίασα ανέφερα ότι οι ανισότητες ε, ξεκινούν, ε, αν ξεκινήσουν από πάρα πολύ νωρίς, από τρυφερή ηλικία, μπορούν να διαρκέσουν πολλά χρόνια και μπορεί να ε, επιβαρυνθούν από τον τρόπο ζωής, από κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους, ε, από κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και έχουν και επιπτώσεις ακόμη και στον προϋπολογισμό. Και μιλάμε για ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις αν ε, δεν δοθεί η απαιτούμενη προσοχή από νωρίς. Έτσι λοιπόν, καθώς το θέμα είναι αυτό πολύ σημαντικό και έχοντας κατά νου ότι το Κοινοβούλιο ήδη ενέκρινε μία σειρά προτάσεων στην έκθεση αυτή, ήθελα να μου πείτε αν η Πολωνική Προεδρία πρόκειται να προσδώσει σημασία ε, στο θέμα αυτό. Τι ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε για να μειώσετε τις ανισότητες στην υγεία. Σας ευχαριστώ. Ähm, λοιπόν, πριν από κάτι εβδομάδες είχαμε επισκεφθεί τον ΕΟΦ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων στο Λονδίνο και εκεί πέρα αναφέρθηκε το θέμα της ανθεκτικότητας στα αντιβιωτικά αφενός και η έλλειψη αντιβιωτικών από την άλλη. Αυτό πρέπει να το ξέρει και το Συμβούλιο. Φαίνεται πως είναι σοβαρό πρόβλημα και θα μας απασχολεί στα επόμενα χρόνια γιατί οι περισσότερες ασθένειες δεν είναι μεταδοτικές αλλά το έχουμε δει και βεβαίως ε, μπορεί αυτά τα φαινόμενα όντως να εξελιχθούν πάρα πολύ επικίνδυνα και χρειαζόμαστε ε, προστασία από μεταδοτικές ασθένειες, πανδημίες ε, και τέτοια πράγματα. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις, αρκετές. Αν θέλετε λοιπόν να απαντήσετε, είμαστε ανυπομονούμε να ακούσουμε τις απαντήσεις σας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, γιατί διαπιστώνω ότι είναι η τελευταία αργάσιμη μέρα σας πριν τις ε, θερινές διακοπές και γνωρίζω ε, τι δύσκολο είναι το έργο σας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος που ασχολείται και με θέματα υγείας. Είναι από, τα, από τους πιο δύσκολους τομείς. Ένα λόγος παραπάνω λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω που ακόμη και την τελευταία εργάσιμη μέρα αφιερώνετε χρόνο για τη συζήτηση μαζί μου. Θα ήθελα πραγματικά εκ βάθους καρδίας να σας προσκαλέσω σε όλες τις διασκέψεις που ανήγγυλα στην προηγούμενη μου ομιλία, στις διασκέψεις των εμπειρογνωμόνων. Γιατί με ενδιαφέρουν οι απόψεις, αλλά θα με ενδιαφέρε και η συμμετοχή σας σε τέτοιου είδους διασκέψεις. Θα σας στείλουμε και προσωπικά προσκλήσεις με τη συγκεκριμένη ημερησία διάταξη και πρόγραμμα των διασκέψεων, ώστε να μπορέσετε να κάνετε το πρόγραμμά σας μετά τις θερινές διακοπές και να κανονίσετε και το δικό σας πρόγραμμα για να μπορέσετε να δώσετε το παρόν και στις διασκέψεις αυτές των εμπειρογνωμόνων. Θα απαντήσω ερωτήσεις όχι με τη σειρά που υπόθηκαν, αλλά ανάλογα με το θέμα που κάλυπταν. Θα ήθελα να πω ότι ε, για μας το θέμα της υγείας ε, είναι εξαιρετικά σημαντικό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, στο, και από, την, ε, από το έργο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το έργο στα Εθνικά Κοινοβούλια και από το επάγγελμά μας όταν είμαστε γιατί ξέρουμε ότι το πιο πολύτιμο αγαθό για τους πολίτες είναι η υγεία. Γι' αυτό και Καταβάλαμε τεράστιες προσπάθειες μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε, ώστε η αίσθηση των συμπολιτών μας να είναι ότι έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στην, στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα υγείας. Και οι διαφορές στην υγεία δεν οφείλονται μόνο στις διαφορές του προσδόκιμου ηλικίας. Ακόμη και στο εσωτερικό της ίδιας χώρας έχουμε ε, σημαντικές διαφορές. Για παράδειγμα, στην ε, Πολωνία υπάρχει διαφορά, ακόμη και μέσα στην ίδια πόλη, στη Βαρσοβία, μεταξύ διαφορετικών συνοικιών, ανάλογα με το αν ε, είναι πιο εύπορη η οικογένεια ή όχι. Και μπορεί να έχει και το προσδόκιμο ηλικία διαφορά ακόμη και 7 χρόνια στις γυναίκες, για παράδειγμα. Οπότε θα πρέπει να αγγίξουμε τους ε, συμπολίτες μας, όχι με απαγορεύσεις, όχι με τιμωρίες, αλλά με πληροφορίες, με διαπαιδαγώγηση. Γιατί δεν φτάνει σωστά η ενημέρωση πολλές φορές μέχρι τους Ευρωπαίους πολίτες. Όσο περισσότερο συνειδητοποιήσουν τα προβλήματα οι πολίτες, τόσο λιγότερες ε, θα είναι και οι δαπάνες υγείας. Όσο περισσότερα γνωρίζουν για την πρόληψη, για τη χρησιμότητα των εμβολίων, αλλά και για τις ε, πολιτικές υγείας και τις εθνικές και τις κοινοτικές, αν γνωρίζει ποιοι, είναι οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί, όσο περισσότερο κατατοπισμένος είναι ο πολίτης, τόσο περισσότερο θα αποφύγει και τις ε, μεταδοτικές νόσους και τις λοιμώδεις νόσους. Μιλούμε σήμερα για προληπτικό εμβολιασμό. Ε, αυτό ε, σε περίπτωση προληπτικού εμβολιασμού δεν έχουμε υποχρεωτικές διατάξεις, είναι συστάσεις, οι προαιρετικές, ε, οι, οι προαιρετικοί εμβολιασμοί. Θα πρέπει όμως να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι ακόμη και αυτοί οι προληπτικοί εμβολιασμοί είναι ασφαλείς και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει διαφάνεια σε όλα τα θεσμικά όργανα ώστε τα προϊόντα που προσφέρουμε, όχι μόνο στα εμβόλια, αλλά και γενικώ τα προϊόντα που προσφέρουμε, τα φάρμακα στους πολίτες, είναι ασφαλή. Θα πρέπει να έχει γίνει σωστό έλεγχος. Η ενημέρωση λοιπόν που αναφέρατε και η ανάγκη σωστή πληροφόρηση των πολιτών είναι κέρια σημασία. Μιλήσετε για τις οδηγίες χρήσεως των φαρμάκων. Το θέμα αυτό πραγματικά είναι επίμαχο. Και γιατί είναι επίμαχο γιατί μερικές φορές είναι τόσο ρευστά τα όρια μεταξύ της διαφήμισης και της ενημέρωσης που σε πολλές χώρες, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες κατά την προσπάθεια αλλαγής οδηγίας ε, έδειξαν επιφυλακτικότητα και δεν τάχθηκαν να φαδών υπέρ της τροποποίησης της οδηγίας. Γι' αυτό και οι χώρες μέλη μετά την αρχική συζήτηση είπαν ότι η νομοθεσία για την παρακολούθηση των ψευδοφαρμάκων, για παράδειγμα, ή παραποιημένων φαρμάκων, είναι πολύ πιο σημαντική από ότι η πληροφόρηση. Εγώ προσωπικά πιστεύω θα πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα αυτό και το φαρμακευτικό πακέτο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την ενημέρωση για τα φάρμακα που δίνονται με συνταγή ε, να τα προωθήσουμε και να λειτουργήσει, να, και για να το επιτύχουμε αυτό στην Πολωνική Προεδρία, προβλέψαμε και διάφορε συναντήσει και επαφέ, αλλά και συγκρότηση ειδική ομάδα εργασία. Για να εξετάσουμε το βελτιωμένο κείμενο τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή το που θα υποβληθεί. Φυσικά στη διάρκεια τη συζήτηση ε, προκύπτει ο βαθμό συμφωνία ή διαφωνία των κρατών μελών με τι διάφορε τροπολογίε Πάντω, Εμεί ευελπιστούμε ότι θα έχουμε αποτελεσματική και επικοδομητική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα με τους ε, εισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές. Τέτοια συνεργασία είναι απαραίτητη για την πρόοδο στη συζήτηση. Σε ό,τι αφορά την ε, δωρεά οργάνων σώματος και τις ε, μεταμοσχεύσεις οργάνων. Στις 5 και 6 Ιουλίου φέτος είχαμε την το πρώτο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας με τη διοργάνωση της Πολωνικής Προεδρίας, υπό την αιγύδα της Πολωνικής Προεδρίας, στο Σόποτ. Και μιλήσαμε και για τις μεταμόσχευσει μεταξύ άλλων. Και διαπιστώσαμε ότι όλο και μεγαλώνουν οι ουρές των ασθενών που περιμένουν μια μεταμόσχευση. Ή επίση είδαμε πόσο στοιχίζει η αιμοκάθαρση, πόσο τεράστια είναι τα έξοδα και πόσο στοιχίζει και στην οικογένεια η επαναφορά αυτού του ασθενούς στην κανονική επαγγελματική, στον κανονικό επαγγελματικό βίο από τη στιγμή που θα σταματήσει την αιμοκάθαρση και θα λάβει μεταμόσχευση ενός νέου οργάνου. Καλό είναι λοιπόν να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι αξίζει να κάνουν δωρεά όργανο σώματος και για τη δική του ζωή και για τη ζωή των συμπολιτών τους. Επίσης μιλήσαμε για τη δωρεά οργάνων από ζωντανούς. Θα πρέπει να τονίσουμε το θέμα της ασφάλειας, της ασφάλειας και για τον δωρητή και για τον ασθενή που θα λάβει το όργανο. Επίσης, ε, επισημάναμε την ανάγκη δικτύου συντονιστών, τη σωστή ανταλλαγή πληροφοριών είπαμε ότι πολύ σημαντικό θέμα θα είναι και η ηλεκτρονική υγεία, η ανταλλαγή πληροφοριών, η ροή πληροφοριών μεταξύ των χωρών μελών για τη δωρεά όργανο Επίσης, πολύ σημαντικό θέμα είναι η θέσπιση κάποιων προδιαγραφών σε ό,τι αφορά τη μεταμόσχευση. Οι Υπουργοί υγεία έδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον για το θέμα αυτό και αισθάνθηκα ιδιαίτερη, ιδιαίτερη γιατί αφιερώσαμε πολύ χρόνο στο θέμα αυτό και τελικά καταλήξαμε και σε κοινή διακήρυξη ότι θα φροντίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υποστηρίξουμε τη μεταμόσχε... τις μεταμοσχεύσεις και τη δωρεά όργανων σώματος. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους ομολόγους μου υπουργού για τη συνεργάσιμη στάση τους. Και η διάσκεψη εμπειρογνωμόνων που στόχο θα έχει μεταξύ άλλων και την ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών, θα γίνει 6 και 7 Οκτωβρίου στο Κατόβιτσε. Φυσικά σας προσκαλώ θερμά και στην ε, διάσκεψη αυτή. Δεν θα γίνει μόνο ανταλλαγή καλών πρακτικών, αλλά θα προετοιμάσουμε και μία συνάντηση για την διαπαιδαγώγηση και παρακολούθηση των εργασιών σε ό,τι αφορά τα βλαστοκύτταρα, ε, τη δωρεά όργανο και αυτά τα θέματα θα ενταχθούν στο πρόγραμμα της διάσκεψης αυτής τέθηκε ένα ερώτημα για τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες και την όσο του Αλτσχάιμερ. Και η προηγούμενη Προεδρία και η Γκρική Προεδρία είχε πολλές εργασίες και στρατηγικές για την καταπολέμηση των νευροεκφυλιστικών παθήσεων, όπως την όσο του Αλτσχάιμερ. Κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να συνεχιστούν αυτές οι εργασίες και πρώτα απ' όλα να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για αυτές τις αρρώσεις που είναι περισσότερο χαρακτηριστικές ε, για την προχωρημένη ηλικία, για την γυραιά ηλικία και πόσο μερικές φορές ε, η πάθηση αυτή περιθωριοποιεί ε, τον ηλικιωμένο. Επίσης θα στηρίξουμε και τις εθνικές πολιτικές υγείας, όπως σας είπα και στην ομιλία μου γιατί έχουμε όλο και μεγαλύτερο αριθμό ηλικιωμένων, αλλά και όλο και μεγαλύτερο αριθμό ηλικιωμένων που νοσούν από τέτοιες νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Ταυτόχρονα θα πρέπει να φροντίσουμε και για αυτούς που δεν είναι άρρωστοι, αλλά φροντίζουν αρρώστους. Να φροντίσουμε για κοινωνική, οικονομική, αλλά και ψυχολογική στήριξη όλων εκείνων των ανθρώπων που ασχολούνται με τη φροντίδα των αρρώστων, αρρώστων από νευροεκφυλιστικές ασθένειες όπως Alzheimer. Θέλουμε να υλοποιήσουμε ένα στόχο που αναφέρεται και στη στρατηγική για το 2020. Και πιστεύω ότι η Πολωνική Προεδρία θα συμβάλλει στην ε, πρόθεση αυτών των στόχων, γιατί πραγματικά θέλουμε να αναβαθμίσουμε την ε, ποιότητα ζωής των ε, ανθρώπων που φροντίζουν αρρώστους ε, με Alzheimer. Επίσης ε, θέλουμε να ασχοληθούμε με τις εγκεφαλοπάθειες, την έγκαιρη διάγνωση, να βελτιώσουμε την πρόσβαση στη φροντίδα αλλά και την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οπότε για να υλοποιήσουμε όλους αυτούς τους στόχους που πολύ σωστά και εσείς ε, συμπεριλάβατε στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική το 2020, θα πρέπει να καταβάλουμε πολλές προσπάθειες. Και μπορεί το βήμα της Πολωνικής Προεδρίας να είναι μικρό, αλλά τουλάχιστον θέλουμε να δώσουμε την όθηση που θα τη συνεχίσουν οι επόμενες Προεδρίες. Και ελπίζω ότι το 2020, όταν θα γίνει ένας απολογισμός στρατηγικής, να είναι θετικός απολογισμός, να έχει σημειωθεί πρόοδος και να μην έχουμε περιοριστεί απλώς σε επίβολες δηλώσεις. τέθηκε μια ερώτηση για τα συστήματα υγείας. Το θέμα αυτό μας απασχόλησε και προς το τέλος της Ουγγρικής Προεδρίας. Οι διαφορές των εθνικών συστημάτων υγείας είναι γνωστές και ορατές. Τις γνωρίζετε, όπως και εγώ. Δεν μπορούν όλοι να προσφέρουν στους ε, ασθενείς, στους πολίτες, συγκεκριμένα ε, όλες τις, ε, μια η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δηλαδή ε, να λαμβάνει κανείς όλες τις υπηρεσίες για τις οποίες καταβάλεις φορές. Δεν είναι η ίδια η ποιότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όλες τις χώρες. Βέβαια ταυτόχρονα διαπιστώνουμε ότι πολύ σημαντικό είναι και η κυριαρχία σε ό,τι την εθνική κυριαρχία σε ό,τι αφορά την οργάνωση του συστήμα, των συστήματων υγείας και αυτό κατοχυρώθηκε και στη συνθήκη της Λισαβόνας. Εμείς ε, στην Πολωνία έχουμε κατοχυρωμένο στο ίδιο το Σύνταγμα την ίση πρόσβαση των πολιτών στην υγεία. Και αυτό το καλάθι των εγγυημένων υπηρεσιών θέλουμε να είναι όσο, πιο, όσο πιο πλούσιο γίνεται. Επίσης ε, δεν θα πρέπει ε, να αποκλείουμε τους ε, ανθρώπους, ε, τους ασθενείς που έχουν σπάνιες νόσους και που η ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη είναι πολύ πιο δαπανηρή. Δεν μπορούμε να περιθωριοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους παραμερίσουμε. Γι' αυτό μίλησα πριν από λίγο για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Γιατί η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι και η στήριξη των συστημάτων υγείας όπου ακριβώς εξαιτία οικονομικών προβλημάτων ορισμένοι άνθρωποι με δαπανηρές ιατροφαρμακευτικές ανάγκες παραμερίζονται. Η ομάδα εργασίας που θα ασχοληθεί με το πρόβλημα αυτό της, των διαφορών στην υγεία και την προσπάθεια εξάλληψης ε, των διαφορών στην υγεία είναι μια ομάδα που θα έχει διευθύνοντα ρόλο σε θέματα υγείας. Τέθηκε μια ερώτηση για τα designer drugs. Ε, ένα νέο είδος ε, ψυχοφαρμάκων, καινούριο φαινόμενο στην Ευρώπη, αλλά πολύ επικίνδυνο. Πρόκειται για διαγερτικά φάρμακα που πολύ συχνά δημιουργούν ε, τέτοιες, ε, τέτοια τοξικότητα που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία. Μερικές φορές ε, η δηλητηρίαση είναι πολύ σοβαρή. Και ενώ για τα γνωστά ε, να γνωρίζουμε ποια είναι τα αποτελέσματα και υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Για αυτά τα designer drugs είναι άγνωστος ο τρόπος συμπεριφοράς μερικές φορές και το μείγμα είναι τέτοιο που τα συμπτώματα είναι άγνωστα και δεν μπορούμε να προσφέρουμε 100% βοήθεια στον ασθενή γιατί ε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να καταπολεμήσουμε τα συμπτώματα. Η Πολωνία τελικά αποφάσισε να απαγορεύσει αυτά τα designer drugs και τον Οκτώβριο ε, είχαμε στην τοξικολογία 260 ε, καταχωρημένους, ε, ενώ πριν από ένα μήνα είχαμε μόνο 4-5 κρούσματα δηλητηρίασης από τέτοια designer drugs. Επίσης, το πρόβλημα έγινε στην παράνομη διανομή και διανομή μέσω του διαδικτύου. Γι' αυτό και τα σύνορα εδώ δεν έχουν νόημα από τη στιγμή που υπάρχουν designer drugs στους γείτονες, ακόμη και τα απαγορεύουμε εμείς, ε, δεν μας ωφελεί σε τίποτα. Γι' αυτό και θα πρέπει από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βρούμε κάποιες κοινές συνταγές για να καταπολεμήσουμε αυτά τα designer drugs που με πολύ ανεύθυνο τρόπο ε, προσφέρουν ορισμένοι ιδιαίτερα στους νέους. Και Είχαμε ένα πρόσφατο παράδειγμα ενός ε, νεαρού εφήβου με πολύ σοβαρά ε, συμπτώματα δηλητηρίασης εξαιτία ε, τέτοιου designer drugs. Υπάρχει ένας κατάλογος ουσιών που απαγορεύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και νομίζω ότι σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να έχουμε μία απρόσκοπτη ροή πληροφοριών για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε αυτά τα, αυτές τις διαγερτικές ε, ε ουσίες και τα ψυχοφάρμακα. Τα θέματα αυτά τα αναφέραμε και στο ΣΟΠΟΤ και είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε να υιοθετήσουμε αποτελεσματικές μεθόδους για να καταπολεμήσουμε αυτά τα νέα ναρκωτικά, αυτά τα designer drugs. Και αυτό θα αποτελέσει προτεραιότητα της Προεδρίας και θα στηρίξουμε την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αξιολογήσει τις εργασίες του Συμβούλου σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή των πληροφοριών, το επίπεδο κινδύνου, σε ό,τι αφορά τις νέες αυτές δραστικές διαγερτικές ουσίες, τα designer drugs, ψυχότροπες και διαγερτικές ουσίες. Σε ό,τι αφορά τώρα το κάπνισμα. Έχουμε μια οδηγία από το 2001 που ισχύει για το κάπνισμα. Σήμερα πραγματικά έχουμε μια επιδημία καπνίσματος και αυτή η επιδημία είναι από τους σημαντικότερους κινδύνους και απειλές του πολιτισμού στον 21ο αιώνα. Σίγουρα εσείς ως ευρωβουλευτές θα ακούσατε και το επιχείρημα ότι αν αυξήσουμε τους έμεσους φόρους κατανάλωσης, γιατί η κατανάλωση μπορεί να οφείλεται και στην τιμή, να εξαρτάται μάλλον από την τιμή των τσιγάρων και ακούστηκε το επιχείρημα ότι αν εμεί αυξήσουμε του έμεσου φόρου κατανάλωση, τότε ουσιαστικά θα, θα ανθίσει το λαθρεμπόριο τσιγάρων ή το παράνομο εμπόριο. Εμείς όμως όσοι ασχολούμαστε με την υγεία γνωρίζουμε ότι και το παράνομο εμπόριο και το λαθρεμπόριο τσιγάρων δεν μπορεί να επηρεάζουν τι πολιτικές μας επιλογές σε θέματα υγείας. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταπολεμήσουμε το κάπνισμα και να συνεργαστούμε και με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας που όπω ξέρετε πολύ γρήγορα, μέσα σε ένα μήνα, κατέθεσε κάποιες μεθόδους αποτελεσματικής καταπολέμησης ε, του λαθρεμπορίου και της παράνομης παρασκευής προϊόντων καπνού. Πάντως για το κάπνισμα περιμένουμε τις εργασίες και τις προτάσεις για την αναθεώρηση της οδηγίας του 2001. Στην προσπάθεια αυτή θα εκμεταλλευτούμε την μέχρι τώρα πείρα των κρατών μελών, αλλά θα αντιμετωπίσουμε και τα νέα προβλήματα της αγοράς και τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Είχαμε συνάντηση με τον Κύπριο Υπουργό Υγεία και μαζί ζητήσαμε από τον Επίτροπο Ντάλι να, να επισπεύσει τις εργασίες για την κατάρτιση οδικού χάρτη για την κατάσταση υγείας και στα πλαίσια αυτού του οδικού χάρτη να συμπεριλάβει και την αναθεώρηση της οδηγίας για το κάπνισμα, για τον καπνό. Βέβαια δεν πρόκειται αυτές οι εργασίες να διεκπαιρεωθούν στη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας. Γι' αυτό και στην αρχή δεν μίλησα μόνο για τις δικές μας προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας, αλλά για τις προτεραιότητες του τρίου των Προεδριών. Ε, θα έχουμε τρεις διαδοχικές προεδρίες που καθορίζουν από κοινού τις προτεραιότητες τους στα πλαίσια του τρίου και ελπίζω ότι τουλάχιστον μέχρι που να τελειώσουν και οι τρεις προεδρίες του τρίου θα έχει ολοκληρωθεί η αναθεώρηση της οδηγίας για το κάπνισμα. Τέθηκε μία ερώτηση για την κοινωνία των πολιτών και αν θα ήταν σκόπιμο να στηρίζουμε περισσότερο την κοινωνία των πολιτών και όχι τους ε, υπαλλήλου των ε, Υπουργείων Υγείας. Και πώς θα πρέπει να επιβραβεύσουμε αυτούς που φροντίζουν για την υγεία σου. Συμφωνώ να επιβραβεύσουμε όσους ε, ασχολούνται και προσέχουν την υγεία τους. Όλοι θα πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι καλό θα ήταν να ζούμε υγιεινά να φροντίζουμε την υγεία μας. Επίσης θα πρέπει να έχουμε επίγνωση και πρόσβαση σε ποιοτικέ υπηρεσίες υγείας όταν αρρωσταίνουμε, αλλά να ξέρει ο καθένας ότι εξαρτάται και από τον ίδιο πόσο θα στοιχήσει, πόσο ακριβά θα στοιχήσει η θεραπεία για όλους. Γιατί μερικές φορές τα χρήματα των συστημάτων υγείας, ο προπολογισμό των συστημάτων υγείας, στο μέτρο που προστίθενται νέες τεχνολογίες, καινοτόμε και νέα φάρμακα, ποτέ δεν θα είναι αρκετά τα χρήματα των προπολογισμών Υγεία, ό,τι και να κάνουμε. Γι' αυτό και θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τον κάθε πολίτη να υπομειστεί την ευθύνη τη υγεία του και τη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ένα συνειδητοποιημένο πολίτη θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη τη υγεία του. Αυτή είναι και η δική μου προσωπική γνώμη, ότι ο θα πρέπει να φροντίζει και για την υγεία του. Σε ό,τι αφορά την κοινωνία των πολιτών, Πολλά μπορούμε να πούμε για το θέμα αυτό. Εμείς έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Έχουμε τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τη δέσμευση πολλών κύκλων, κέντρων, Ινστιτούτων, πολλών ενώσεων που προωθούν τον υγιεινό τρόπο διαβίωσης προσπάθεια σωστής διαπαιδαγώγησης των νέων γενιών και κυρίω των παιδιών από μικρή ηλικία να μπουν τα σωστά θεμέλια για την υγεία. Αυτό είναι ανεκτήμητο πραγματικά. Να μπουν από την αρχή στέρε βάσεις για μια σωστή διαπαιδαγώγηση στα θέματα υγείας υγιεινής ζωή. Και μία ακόμη τελευταία ερώτηση. Νομίζω ήταν δική σας, κύριε Ευρωβουλευτά, για τα τρόφιμα για τα νέα τρόφιμα, τα novel foods. Υπάρχει ε, νομοθετική ρυθμισή ευρωπαϊκή με βάση τον κανονισμό για τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά των τροφίμων και όπως θυμόμαστε όλοι, τον ε, Ιανουάριο του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο μία πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού για τα νέα τρόφιμα. Η Πολωνία τάχθηκε υπέρ της αναθεώρησης. Η ρύθμιση για την ανατεχνολογία τελικά μεταφέρθηκε σε ένα σχέδιο κανονισμού σε σχέση με την ενημέρωση των καταναλωτών για θέματα, των, για θέματα τροφίμων. Συνεχίζονται ακόμη οι εργασίες για τον κανονισμό αυτό. Η Ουγγρική Προεδρία είχε προτείνει λοιπόν να περιληφθεί στην ε, οδηγία για τα νέα τρόφιμα, γιατί τρόφιμα που περιλαμβάνουν ή αποτελούνται από νανοηλικά θα πρέπει να υπόκειται στην οδηγία αυτή. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά την υποβολή του νέου σχεδίου κανονισμού για τα νέα τρόφιμα. Δεν γνωρίζουμε το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε δεν μπορώ να προκαθορίσω και να προεξοφλήσω πότε θα ασχοληθούμε εμείς με το θέμα αυτό. Πάντως, ένα πράγμα μπορώ να εγγυηθώ, ότι μόλις λάβουμε τις πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ασχοληθούμε προσεκτικά με το θέμα αυτό και θα εργαστούμε φυσικά άοκνα για να το προωθήσουμε. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι τα κάλυψα όλα. Αν διέχει κάτι. Ναι, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου. Νομίζω πως ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση με πάρα πολλά θέματα. Ο κύριος Σάρης Βόλσκι μας παρακολούθησε και αυτό στο τελευταίο μέρος. Ενδιαφέρεται και αυτός για την υγεία, εννοείται, όπως και για πολλά άλλα πράγματα σε αυτό το κοινοβούλιο. Νομίζω λοιπόν πως απαντήσατε πολύ σωστά. Βλέπουμε πως ε, σας απασχολεί το θέμα της υγείας ε, και βεβαίως ε, είναι σοβαρό θέμα και για την Πολωνική Προεδρία. Αναφέρατε διάφορες διασκέψεις για την Προεδρία και απευθύνατε και πρόσκληση στα μέλη εδώ του Κοινοβουλίου. Οπωσδήποτε θα συνεργαστούμε καλά, σας διαβεβαιώ γι' αυτό, επικοδομητικά. Ελπίζουμε να έχετε καλή επιτυχία, γιατί πράγματι ο κόσμος περιμένει η Ευρώπη να παίξει και εδώ πέρα ένα χρήσιμο ρόλο στην προσπάθεια να ζει κανείς υγιεινά. Και όταν ταξιδεύει κανεί σε άλλη χώρα, όταν δουλεύει σε άλλη χώρα, όταν πάει διακοπέ, Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχουν διάφορα έργα που προετοιμάζονται. Καλή επιτυχία λοιπόν και θα τα ξαναπούμε είτε στο Στρασβούργο είτε εδώ στην Επιτροπή μας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και ευχαριστώ που ήρθατε. Bardzo Σας ευχαριστώ θερμά. Και θα ήθελα να απευθώ φυσικά σε όλους τους ευρωβουλευτές. Όταν ήρθα, ο μόνος μου φόβος ήταν ότι θα μιλάω σε άδεια αίθουσα. Γιατί είμαι η τελευταία υπουργό που προβλεπόταν να παρουσιάσει τις πολωνικές προτεραιότητες. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά που έστω και αυτή την τελευταία εργάσιμη μέρα δώσατε το παρόν και σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις που μου έδωσαν τροφή για σκέψη και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για μια πολύ σημαντική δήλωση που κάνατε. Είπατε ότι εσείς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ε, άνθρωποι που δεν αρνούνται την βοήθεια, δεν αρνούνται τη συνεργασία και το επόμενο εξάμεινο θα συνεργαστούμε ε, στενά και επικοδομητικά για την πρόθεση της υγείας στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και το επανειδήν.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 So, Έχουμε τώρα δύο θέματα, δύο προφορικές ερωτήσεις. Ε, μία του Πέτερ Λίζε, θα συζητηθεί τώρα. Το θέμα δηλαδή που αφορά. Α, ah, Α, και η δεύτερη είναι δικιά σου, Λίντα. Όσον αφορά μια οδηγία για οικολογικό σχεδιασμό και ο Πέτερ Λίζα πιθανή σχέση κινητού τηλεφώνου και αυξημένου κινδύνου καρκίνου. Εγώ μόλις μίλησα με τον Πίτερ και λέει να τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτα να δούμε την εφαρμογή και μετά το άλλο, γιατί εγώ πρέπει να προλάβω και το τρένο μου. Δεν θα αργήσουμε λοιπόν. Ας δούμε τώρα τα της εφαρμογής. Ο Πίτερ δεν έχει πρόβλημα. Tak. Przechodzimy do punktu 24. Προχωρούμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, στο 24ο. Έχουμε και την e, Εθνική Εορτή της Γαλλίας σήμερα. Δεν βλέπω κανένα Γάλλο. Για να του ευχηθώ. Θα ήθελα πάντως e, να ευχηθώ σε όλους τους Γάλλους, ευρωβουλευτές, βοηθούς, υπαλλήλου. να τους συγχαρώ για την εθνική τους ε, γιορτή. Προχωράμε στο επόμενο σημείο λοιπόν της ημερήσιας διάταξης, την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για το Περιβάλλον και την οδηγία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την οδηγία ΡΟΣ. który jest reprezentantem komisji. Proszę bardzo, panie Brekle. Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρακαλώ. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ. Λέγομαι Πιέλ Χάντσεν από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ περιβάλλοντος και χημικών προϊόντων. Είμαι εδώ για θέματα που αφορούν το REACH. Σημείο 3. Αρμόδιος είναι ο κύριος Μπράκλαντ που έπρεπε να είναι εδώ για να απαντήσει στην ε- έκθεση, στην προφορική ερώτηση της κυρίας Μακάβαν. Τη σχέση της οδηγίας ΡΟΣ με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι εδώ ο κύριος Μπράκλαντ. Κύριε Μπράκλαντ, μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτηση της κυρίας Μακάβαν. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Η Κομισιόν ε, γνωρίζει ότι ο περιορισμός ε, των επικίνδυνων ουσιών ε, στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό κανονισμό για τι επικίνδυνε ουσίε θέτει πάρα πολύ ψηλά πρότυπα στην περιβαλλοντική προστασία. Η εφαρμογή είναι το σημαντικότερο. Έτσι λοιπόν συμφωνεί η Κομισιόν ότι είναι μέγιστη σημασία για τι μικρέ και μισέ επιχειρήσει ε, να λαβούν τη μέγιστη υποστήριξη τη διοικητική. Εμεί σκοπεύουμε να υποστηρίξουμε την εφαρμογή τη οδηγία, ε, να θέσουμε προτεραιότητα στο έργο για την ε, εξαίρεση και επίσης ε, να απαντούμε ε, στις εταιρείε όταν ε, μας θέτουν αποσοφιστικές ερωτήσεις. Επίσης είμαστε σε στενή επαφή με τους προσώπους της βιομηχανίας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε τακτική βάση και η παραγωγή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ενημερώνονται για τις απαιτήσει ε, και από ό,τι κατάλαβε, κύριε Μακβάν, ήρθε και σε επαφή, το γραφείο της ήρθε σε επαφή με την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Περιβάλλοντος. Επίσης, υπάρχουν και κάποια τεχνικά ε, θέματα. η οδηγία ΡΟΣ περιλαμβάνει σημαντικές ε, διατάξεις για τις εξαιρέσεις από την απαγόρευση των ουσιών αυτών, γιατί υπάρχει δυσκολία εφαρμογή στην πράξη. Έτσι λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, δηλαδή αν υπάρχει κάποια αμφιβολία για το τι σημαίνει η διάταξη, υπάρχει δυνατότητα εξαίρεση. Η εξαίρεση βασίζεται ε, στην εφαρμογή από την ηλεκτρονική βιομηχανία και αναφέρεται σε συγκεκριμένα ε, υλικά και πολλέ φορέ ο παραγωγό θα ξέρει καλύτερα για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Έτσι λοιπόν ε, ε, αυτό αφορά ε, τους παραγωγούς και αν δείτε την, οδηγία, την ανδιατύπωση της οδηγίας που δημοσιεύτηκε και πάλι Ιουλίου 2011 θα δείτε ότι στον κατάλογο των εξαιρέσεων στο παράρτημα 3 πολλές φορές έχετε προσδιορισμό πολύ συγκεκριμένων προϊόντων. Πάντως επειδή είναι πολύ προκατατεχνικά τεχνικά ζητήματα και υπάρχει αμφισημία, υπάρχει αμφισημία σε σχέση με το πεδίο εφαρμογή των εξαιρέσεων κυρίως όταν διαφέρει πάρα πολύ χρήση του προϊόντο σε σχέση με την αρχική εφαρμογή. Παραδείγματο χάρη, αναφερόμαστε εδώ σε έλαπε που χρησιμοποιούνται στα αεροδρόμια και ε, έτσι λοιπόν, αν μόνο το δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί για την πρακτική εξαίρεση, τότε εμεί υποστηρίζουμε την εξαίρεση στην περίπτωση αυτή και οι ε, ετούντε ακολουθούν ε, την συμβουλή τη Κομισιόν ότι θα ζητήσει ο παραγωγό για πιο συγκεκριμένη εξαίρεση εξαίρεση για το προϊόν. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκη η οδηγία στις ε, συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις. Ε, ακόμη και ο Σύμβουλος κομισιών δεν μπορούσε να δώσει συγκεκριμένη απάντηση για το πεδίο εφαρμογή του ορισμού, αλλά τελικά βρήκαμε μια πρακτική λύση μέσω της εξαίρεσης για την οποία, την οποία θα ζητήσει εν λόγω εταιρεία. Ευχαριστώ κυρία Μαγκάβαν για συμπληρωματική. Ναι. Ε, είναι τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά για να ξέρουν και οι συνάδελφοι. Το θέμα είναι όταν δεν ξέρει μια εταιρεία εάν ένα προϊόν της καλύπτεται από μια εξαίρεση για την οδηγία ΡΟΣ. Και το θέμα είναι ότι κανείς δεν μπορεί να του δώσει απάντηση, ούτε η Κομισιόν, από το, για το αν εξαιρείται το προϊόν τους ή όχι, ούτε το, το Οικολογικό Ινστιτούτο που εφαρμόζει για την Κομισιόν την οδηγία. Οπότε εμείς ως νομοθέτες ε, να ξέρουμε ε, την νομοθεσία και μου είπαν πως η εταιρεία είναι μια μικρή εταιρεία και τις είπαν να βρουν ένα δικηγόρο και να τα βρει αυτός και αλλιώς θα αναλάβουν τον κίνδυνο να αντιμετωπίσουν μηνύσεις. Ε, δεν είναι πράγματα αυτά, πρέπει να είναι σαφές ποιον καλύπτει ο νόμος, ποια προϊόντα κτλ. Επίσης, ε, το Οικολογικό Ινστιτούτο είπαν πως δεν μπορούσαν να βοηθήσουν με μονομένες εταιρείε, δεν τους πλήρωνε γι' αυτό η Κομισιόν. Οπότε ποιος μπορούσε να βοηθήσει αυτή την ε, οδηγία. Οπότε δεν βλέπω να το λύνουμε σήμερα, αλλά είναι ικανοποιητικό. Και εγώ δεν θεωρώ ότι τους απαντάω σωστά ως Ευρωβουλευτής να τους πω «Α, απομισθείτε εσείς το ρίσκο και βρείτε μόνοι σας αν σας καλύπτει ή όχι». Ε, δεν είναι έτσι. Εξευθελιζόμαστε στα μάτια του κοινού. Αν δεν ξέρουμε εμείς ε, αν καλύπτεται κάτι ή όχι, πού να ξέρουν οι άλλοι. Είναι μια μικρή εταιρεία που θέλει να ξέρει αν όχι καλύπτεται από αυτό ή όχι. Θέλετε να απαντήσετε. Συμφωνώ και εγώ πλήρως και εγώ δεν ξέρω. Οι εταιρείε πράγματι πρέπει να ξέρουν ε, τι ισχύει. Ήρθαμε σε διαβουλεύσεις ε, με Καταναλωτέ, ε, Υπάρχει πρόβλημα με τις μικρομεσαίε επιχειρήσει να τις βρουν. Προσπαθούμε να βρούμε μια θετική λύση μέσω τη εξαίρεση. Ε, πρέπει να βρουν τι, τι γίνεται μόνοι τους. Πράγματι δεν είναι ιδεώδες από πλευράς ε, νομοθεσία και καταλαβαίνω πως το ίδιο, το ίδιο πράγμα κάνουν και άλλες εταιρείε. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do Περνάμε στην επόμενη ερώτηση της κυρίας Κάντεμπαχ. Η κυρία Κάντεμπαχ έθεσε ερώτηση για τα προβλήματα εφαρμογής στα κράτη-μέλη. Αυτό έλεγε τουλάχιστον στην προφορική ερώτηση. Ποιος είναι αρμόδιος απαντήσει. Και πάλι ο κ. Σάκλαντ είναι αρμόδιο να απαντήσει για τα προβλήματα εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Ε, Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε με τον ε, επικεφαλή ε, των νομικών υποθέσεων. Η ερώτηση είναι αν υπάρχει μια μελέτη σχετικά με τον γιατί τα κράτη-μέλη έχουν πρόβλημα να εφαρμόσουν το δίκαιο του περιβάλλοντος και τι κάνει η Κομισιόν. Από όσο γνωρίζω δεν έχει γίνει μια συνολική μελέτη από την Κομισιόν για το θέμα αυτό. Μπορεί να βρείτε κάποια γενικά σχόλια στη Λευκή Βιβλό για την διακυβέρνηση, για τη γενική εφαρμογή της Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Από όσο γνωρίζω θα έλεγα ότι υπάρχουν πολλά κριτήρια που εξηγούν τη δύσκολη εφαρμογή Καταρχήν, η περιβαλλοντική νομοθεσία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε οδηγίε και αυτό νομίζει ότι ε, σημαίνει ότι έχουμε μεταφορά στην εθνική νομοθεσία από τα κράτη-μέλη και από τι ε, αρχέ τη τοπική αυτοδιοίκηση και επίση υπάρχει και το πρόβλημα του ότι ε, δεν συνάδει τελικά η εσωτερική νομοθεσία με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Επίση, υπάρχει μεγάλη αποκέντρωση και η εφαρμογή δεν γίνεται σε εθνικό επίπεδο ούτε καν σε επίπεδο τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά μπορεί να γίνει γίνεται σε επίπεδο Μιλάμε επίσης για θετικές υποχρεώσεις. Πρέπει να οικοδομηθούν ε, πράγματα. Έτσι λοιπόν υπάρχει μεγάλος ε, συσχετισμό με τις υποδομές και χρειάζονται και χρήματα. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι αν ε, συγκρίνουμε το περιβαλλοντικό δίκαιο με την ενιαία αγορά που έχουμε περισσότερες αρνητικές υποχρεώσει, δηλαδή να μην κάνετε πράγματα εδώ, ε, περισσότερο ζητείτε να δημιουργηθούν υποδομές, ε, το χάρη μέσα σε δύο εβδομάδε ε, δεν μπορούν ε, να ε, δημιουργηθούν κάποιες μονάδες για την επεξεργασία των λιμάτων, παραδείγματο χάρη. Δέκα χρόνια χρειαστήκαμε στις Βρυξέλλες ε, για να οικοδομήσουμε το εργοστάσιο. Επίσης, ε, η περιβαλλοντική νομοθεσία ήταν η πρώτη που χρησιμοποίησε, που, συγγνώμη, που δημιούργησε περιβαλλοντικέ υποχρεώσει. Για πολλά κράτη-μέλη, λοιπόν, αυτή η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσουν από το μηδέν. Γι' αυτό είναι τόσο πολύπλοκο το θέμα. Υπάρχει και ένα γενικό πρόβλημα που είναι η έλλειψη ικανοτήτων στι εθνικέ δικασίες Πολλέ φορέ δεν υπάρχουν επαρκεί πόροι ή επαρκεί γνώσει για να τεθεί σε εφαρμογή το περιβαλλοντικό δίκαιο. Τη Ευρωπαϊκή Ένωση Έχουμε λοιπόν μια ευρία γκάμα προβλημάτων και ο Επιτροπή μου θα ήθελε να κάνει μια ανακοίνωση για την εφαρμογή τη περιβαλλοντική νομοθεσία. Πιστεύει ότι η εφαρμογή μαζί με την βιοπικιλότητα και την αποδοτικότητα των πόρων αποτελούν ύψε προτεραιότητε. Έτσι λοιπόν θα παρουσιάσει ένα εγγραφό το οποίο θα αποτελεί μια διάγνωση της αποτυχίας εφαρμογής και ορισμένες συστάσεις. Είχαμε για αυτό το θέμα μια διασκέψη πρόσφατα, 15 Ιουνίου, είχαμε ένα καταιγισμό ιδεών, συμμετείχαν και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το τι μπορεί να γίνει. Καταρχήν, ε, μια επιλογή είναι να αυξήσουμε την ενημέρωση των πολιτών και μια άλλη δυνατότητα είναι να, να βελτιώσουμε τη διακυβέρνηση ε, στα κράτη-μέλη. Τώρα, για να, να αναφέρομαι στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνηση, πρέπει να υπάρχει σύνδεσμο μεταξύ του, επίση πρέπει να υπάρχει σύνδεσμο με τη χρηματοδότηση και σύνδεσμο με τη δικαιοσύνη. Δεν ε, υπάρχει τέτοια εγγύηση σύνδεσμο με τη δικαιοσύνη στα κράτη-μέλη. Εν τω μεταξύ προσπαθούμε να, είμαστε, να συνεργαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο με τα κράτη-μέλη και θα αναφέρω ένα παράδειγμα στο παρελθόν όταν υιοθετήθηκε η οδηγία από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο τα κράτη-μέλη θα αφήνονταν ε, κατά μέρου και κατά κατόπιν ε, θα άρχιζε η Κομισιόν να λέει δεν έχετε μεταφέρει στο ιστορικό δίκαιο και θα αρχίζουν διαδικασίε σε παραβάση. Τώρα, εμεί προσπαθούμε να αναλάβουμε προληπτική δράση στη δική μου ε, διεύθυνση. Προσπαθούμε να στέλνουμε και ένα checklist ε, σε σχέση με τα προβλήματα για τη μεταφορά της νομοθεσίας στο ιστορικό δίκαιο. Προσπαθούμε να ανταλλάσσουμε τις βέλτιστες πρακτικές και τα διδάγματα Πολλά λοιπόν μπορούν να γίνουν για τη βελτίωση της εφαρμογής, ε, διαφορετικές ιδέες θα παρουσιαστούν από τον Επίτροπό μου στα τέλη του έτους, αλλά υπάρχουν και κάποιες πιο πρακτικές ιδέες για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη πιο σωστά να μεταφέρουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στο εθνικό τους δίκαιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μήπως η κυρία Κάντεμπαχ θέλει το λόγο. Να σας ευχαριστήσω για αυτά που είπατε. Νομίζω πως χρειάζεται μια συγκριτική μελέτη, γιατί δεν έχει νόημα η ωραία νομοθεσία όταν διαπιστώνουμε πως ε, δεν εφαρμόζεται σε μια σειρά κρατών μελών. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια βάση για να ξέρουμε πως ε, θα υπάρχει νομίζω η σωστή υποστήριξη. Γιατί βλέπουμε κομματάκια ενό παζλ και αντιδρούμε σε αυτά, αλλά δεν έχουμε μια ε, γενική εικόνα και θα μπορούσε να μα το δώσει μια μελέτη. Μια άλλη παράκληση. Θα ήθελα την απάντηση στην ερώτηση παριθμών 5 για τις επιθεωρήσεις ε, στην Ιρλανδία. Εάν θα μπορούσατε να την απαντήσετε, ευχαριστώ. Tak, pani. Pytanie Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την ε, εξόριξη τύρφης. Ήταν μια ερώτηση που την έθεσε αρχικά η κυρία Childers και την αναπληρώνει εδώ η κυρία Κάτεμπαχ. Μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό ερώτηση για την εξόριξη τύρκη στην Ιρλανδία. Ναι, ευχαριστώ. Είμαι υπεύθυνο και εγώ για είναι διευθυντή που υπεύθυνη για το θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν, η ερώτηση αφορά την εξόριξη τύρφη στην Ιρλανδία και το ότι οι τυρφώνες ε, βρίσκονται σε ένα οικοσύστημα και παρά την ευρωπαϊκή προστασία ε, εξακολουθεί να υπάρχει τέτοια δραστηριότητα εξόρεξης τύρφης. Παρακολουθούμε πολύ στενά αυτή την κατάσταση. Έχουμε ξεκινήσει διαδικασία παραβάση κατά της Ιρλανδίας. Έχουμε στείλει επίσημη επιστολή στα τέλη του Ιανουαρίου του 2011. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η νέα κυβέρνηση είχε κάνει σημαντική προσπάθεια για να επιλύσει το ζήτημα, για να το θέσει ως προτεραιότητα το ζήτημα δημιουργώντας παραδείγματος χάρη ένα συμβούλιο για την τύρφη και προσφέροντας αποζημίωση σε όσους κατέχουν ε, λιβάδια τύρφης ε, και ασκώντας διώξεις όσους καταστρέφουν ε, το οικοσύστημα, τον οικότοπο. Και, όμως στο στάδιο αυτό πιστεύουμε ότι πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα από την Ιρλανδική, Ιρλανδική κυβέρνηση. Δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από την εφαρμογή των μέτρων ε, από την Ιρλανδική κυβέρνηση, από τις Ιρλανδικές αρχές. Γι' αυτό η Κομισιόν ε, υιοθέτησε τη λογική είναι γνώμη φέτος 26 Ιουνίου και η προθεσμία για την απάντηση είναι η 16 Ιουλίου για τις Ιρλανδικές αρχές. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα είναι ένα μήνα η προθεσμία αντί για δύο μήνες. Και έτσι λοιπόν ε, η Κομισιόν μπορεί να μετακινηθεί νωρίτερα στο επόμενο στάδιο αν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Προ στιγμή οι πληροφορίε που έχουμε είναι ότι οι καταστροφές ε, του 56ου, της 56 περιοχής έχουν ε, σταματήσει, αλλά έχουμε και ακόμα 200 τέτοιες τοποθεσίες όπου συμβαίνει τέτοια δραστηριότητα και όπως σας είπα θα παρακολουθούμε πολύ στενά πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Αρκεί η απάντηση, έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε τον Διευθυντή, τον κύριο Μπράκλαντ, που ήρθε για να απαντήσει. Ολοκληρώνουμε το σημείο αυτό. Και όσες προφορικές ερωτήσεις έμειναν λόγω απουσίας ευρωβουλευτών, θα αναβληθούν για την επόμενη συνεδρίαση. Πολύ ευχαριστώ τις αναλάβω εγώ για, για το ρίτσο, ας πούμε, αν σας ε, εξυπηρετεί. Αν εμ, μπήκαν στον κόπο να έρθουν μέχρι εδώ εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορούμε κάλλιστα να ακούσουμε τις απαντήσεις, αναλάβω εγώ τις ερωτήσεις. Mm, Ήταν η ερώτηση του κυρίου Λίζε. Αν συμφωνούν οι συνάδελφοι, θα ήθελα να παρακαλέσω την Κομισιόν να πει κάτι για τα κινητά τηλέφωνα. Πριν μετά δεν με ενδιαφέρει, απλά το συνεννοήθηκα με τη Λίντα Μακάβαν γιατί πρέπει μετά όλοι να φύγουμε, να πάμε στη χώρα μας. Καλώς. Προτείνω μια σολομόντια λύση. Να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Λίζε και μετά μπορούμε, αν θέλετε, να επανέλθουμε στα προηγούμενα θέματα. Αν ε, έχει την καλοσύνη να παραμείνει λίγο ακόμη ο διευθυντής ε, Χάνσεν. Κύριε Λίζα, προφορική ερώτηση σε ό,τι αφορά την πιθανή σχέση μεταξύ χρήση κινητού τηλεφώνου και αυξημένου κινδύνου καρκίνου. Ο κύριο Βίλεμ Πένιγκ είναι πρόσωπος, ή η κυρια μάλλον. Κυρία ή κύριο κύριος Βίλεν Πένινγκ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο, κύριε Διευθυντά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω στο ερώτημα του κυρίου Λίζε και του κυρίου Ζέμπερ. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα για εμάς, γιατί, ε, ξέρετε, 31 Μαΐου 2011 η Διεθνής Υπηρεσία Έρευνας ε, Καρκίνου, που είναι φορέας του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, κατέταξε τις ε, ε και τα ηλεκτρονικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία των κινητών τηλεφώνων ως πιθανός καρκινογόνα. Για να γίνει αυτό δεν έγινε μελέτη, όπως αναφέρεται στην αρχική ερώτηση των κυρίων βουλευτών, αλλά μελέτησαν ε, τα υπάρχοντα επιστημονικά στοιχεία σε μια δομημένη διαδικασία αξιολόγησης ε, υπαρχόντων ε, στοιχείων από ομάδες ειδικών. Τελική κατάταξη μετά από συζητήσεις δύο εβδομάδων κατέληξε σε αυξημένο κίνδυνο γλιωμάτων σε κάποιες ε, επιδημιολογικές μελέτες σε ε, πολύ συχνούς χρήστες ε, των κινητών. Υπάρχει λοιπόν, όπως είπαμε, περιορισμένος κίνδυνος καρκινογένεσης από τα κινητά ε, τηλέφωνα. Οι συνάδελφοί μου ήταν παρόντες σε αυτές τις συζητήσεις και μπορούμε να πούμε πως ε, η κρίση αυτή αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής διαφωνίας και υπάρχει και η γνώμη της μειοψηφίας όπως ξέρετε. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε πως τα δεδομένα αυτά θεωρήθηκαν ανεπαρκή για να βγουν συμπεράσματα για οποιονδήποτε άλλο τύπο καρκίνου και σενάριο έκθεσης. Θέλω να το τονίσω αυτό, ειδικά όσον αφορά πηγές έκθεσης μεταξύ των οποίων και κεραίες με τις οποίες συνδέονται τα κινητά τηλέφωνα. Και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Συμφώνω προς τη συνθήκη, τα κράτη-μέλη τα οποία είναι υπεύθυνα για την προστασία του κοινού από πιθανές επιπτώσεις ε, ε, από ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα, οπότε μόνο τα κράτη-μέλη έχουν άμεσα μέσα στην διάθεσή τους για να μειώσουν την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Στο πλαίσιο αυτό, Πρέπει να σας πούμε πως το 1999 η Κομισιόν πρότεινε όρια έκθεσης και κατά οποία είχε ζητήσει το Συμβούλιο για να συστήσουμε κάποια όρια έκθεσης ε, του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ειδικά αυτά που δημιουργούνται από τα κινητά τηλέφωνα το καθήκον εφαρμογής αυτής της μη δεσμευτική ε, σύστασης, όπως είναι όλες οι συστάσεις βεβαίως, ε, είναι καθήκον των κρατών μελών. Τι κάνει τώρα η Κομισιόν. Η Κομισιόν οπωσδήποτε δεν κάθεται και λέει κάντε το καθήκον σας. Παρακολουθεί συνεχώς τα ευρήματα της ε, επιστήμης στον τομέα αυτών με, βα... με τη βοήθεια μιας ανεξάρτητης επιστημονικής επιτροπής αξιολόγησης των κινδύνων στην υγεία. Στόχος είναι να αξιολογηθεί η εγκυρότητα των ορίων που είχαμε ορίσει τότε στην σύσταση αυτή του 1999 υπαριθμών 519. Η τελευταία γνωμοδότηση για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που υιοθετήθηκε είναι του 2009 και δεν έδινε τότε ένα σκεπτικό για τα τροποποιημένα όρια έκθεσης που υπάρχουν στη σύσταση του Συμβουλίου. Τώρα η Κομισιόν ήδη και πριν από την υιοθέτηση στις 31 ε, Μαΐου 2011 σκόπευε να οργανώσει μια επιστημονική συζήτηση, μια διάσκεψη για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τη δημόσια υγεία. Και αυτό είχε ήδη προγραμματιστεί για τις 16 και 17 Νοεμβρίου. Στο συνέδριο αυτό θα δούμε που υπάρχει επιστημονική συνένεση για τις ε, πιθανές συνέπειες για την υγεία των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και να προτείνουμε μια στρατηγική για να δούμε τα επιστημονικά κενά που παραμένουν. Στο τέλος του 2011, μετά την διάσκεψη και λαμβάνοντας υπόψη ε, το αποτέλεσμα, θα υποβάλουμε νέο αίτημα στην Επιστημονική Επιτροπή για να επικαιροποιήσει τη γνωμοδότηση αυτή για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία βασισμένα στα τελευταία στοιχεία για να ανακαλύψουμε όλα τα ζητήματα υγείας και όχι μόνο τον καρκίνο. Υπάρχουν επίσης άλλα τρία στοιχεία που απασχολούν αυτή τη στιγμή την Κομισιόν. Το πρώτον, τη βάση της ε, έκθεσης αυτής και την ε, επάρκεια, όπως σας είπα, της ίστασης 1999 και το εάν χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να δούμε εάν ε, χρειάζεται να καλυφθούν και κάποια άλλα τα οποία δεν είναι ακόμα πλήρως κατανοητά. Δεύτερον, χρηματοδοτήσαμε και θα χρηματοδοτήσουμε έρευνα μέσω του προγράμματος ε, πλαισίου για να κλείσουμε τα γενιά ε, κενά που υπάρχουν στην επιστημονική γνώση για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Και τέλος θα έχουμε έναν διάλογο των ενδιαφερομένων για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και την υγεία για να βρούμε τα ειδικά ζητήματα τα οποία μας ε, θέτουν οι ομάδες πίεσης για να αντιληφθούμε καλύτερα την κατάσταση και κοιτάμε ήδη και τώρα το πώς μπορούμε να ενημερώσουμε καλύτερα το κοινό για την ε, πολιτική την οποία ακολουθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σιλίζε. Ευχαριστώ, ζητώ συγγνώμη γιατί πρέπει να ξαναφύγω αμέσω γιατί φεύγει και το τρένο. Οπότε δεν υπάρχει καμία ερώτηση, δεν θα ήταν σωστό γιατί δεν θα ακούσω την απάντηση. Μία παράκληση μόνο προς την Κομισιόν. Να το πάρει σε σοβαρά αυτό το θέμα και σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία έχουμε ένα πρόβλημα και αν διαφωνούν οι επιστήμονες υπάρχει ε, σχέση, γιατί το ζήτημα είναι η διαφωνία, το αντικείμενο της διαφωνίας είναι ε, πόσο αιτιώδης, ε, πόσο ισχυρός είναι ο συσχετισμός μεταξύ της ακνοβολίας και της ασθένειας. Να θυμηθούμε τι είχαμε κάνει στο παρελθόν. Εξάλλου έχουμε και το θέμα της διοξίνης που ξέρουμε πως είναι επικίνδυνη και το ζήτημα πάλι είναι οι ποσότητες ακριβώς. Ε, αν και κάποιοι επιστήμονες λένε πως δεν υπάρχουν ε, βλάβες. Οπότε εδώ πέρα υπάρχει σχέση μεταξύ κινητών τηλεφώνων και όγκων. Το... Η έκταση είναι το θέμα, αλλά νομίζω πως το θέμα αξίζει να είναι ξανά στην ημερήσια διάταξη για είμαι περισσότερους συναδέλφους παρόντες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Πένινγκ για τις διευκρινήσεις που μας έδωσε. Και επανέρχομαι στο προηγούμενο σημείο, το 24. Υπάρχει όμως ένα διαδικαστικό ζήτημα εδώ, γιατί την ερώ... τις ερωτήσεις για το ρίτς τις έθεσαν η κυρία Γκροστέτ και η κυρία Γκίρλινγκ που απουσιάζουν. Δεν ξέρω αν ο κύριος Ντέιβις θέλει το λόγο αλλά ούτως ή άλλως πρέπει να το αναβάλουμε όταν θα είναι παρούσες οι συντάκτηρες ερώτησης, δεν ξέρω. Ε, η απουσία της κυρίας Γκροστέτ φυσικά είναι δικαιολογημένη, είναι η γαλλική εθνική εορτή. Νομίζω ότι καλύτερα να επανέλθουμε στο θέμα αυτό της στην επόμενη συνεδρίαση. Απ' την άλλη είναι παρόν ο διευθυντής Χάνσεν που ήρθε επί τούτου για να απαντήσει σε ερωτήσει. Εντάξει, ακούσουμε κάποια σχόλια τώρα, στοιχεία και να επανέλθουμε όταν θα είναι παρούσα και η συντάκτηρα της ερώτησης, κυρία Γκροστέτ. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν θέλω να σκίσω πίεση. Απλά Κομισιόν ήρθε εδώ στη συνεδρίαση και δεν έχει την, ε, τη δυνατότητα να συνεισφέρει. Είναι πάντοτε δύσκολο με τις συνεδριάσεις, ε, Πρόεδρε. Είναι ιδιαίτερα πολύτιμες, αλλά πολύ συχνά, ξέρετε, τυχαίνει να είναι στο τέλος ε, της συνεδρίασης σε τέτοιες ημέρες Σας ευχαριστούμε. Νομίζω ότι είναι συνετό να αναβάλουμε το σημείο αυτό για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Κύριε Διευθυντά, θα πρέπει να το ανα... αναβάλουμε για την επόμενη φορά.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 Écoutez, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σημείο 26. Προτείνω ένα τέταρτο διακοπή. Και θα επανέλθουμε σε ένα τέταρτο εφόσον έχει στο μεταξύ καταθάσει και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Euh, euh, Δεν χρειάζεται καν να διακόψουμε. Γιατί ήρθε στο μεταξύ και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Πολ Χάτσον. Άρα Περνάμε στο σημείο 10. 26 σχέδια θελοντική συμφωνία που θα συναθεί στο πλαίσιο τη οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό με στόχο τη βελτίωση τη ενεργειακή απόδοση των σύνθετων ψηφιακών αποκωδικοποιητών και την εκτίμηση των επιπτώσεών του. Παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας κάνει ο κύριος Πολ Χάτσον, Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα. Κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και καλησπέρα σας. Αυτή είναι μια εκούσια συμφωνία στην οποία ερχόμαστε στην νόμη τη ε, οδηγίας ε, για τον οικολογικό συνδυασμό. Αυτή η οδηγία επιτρέπει να αναγνωρίζονται εκούσες συμφωνίε σε ορισμένε περιπτώσεις ε, ως μια εναλλακτική ισχύουσα έναντι του κανονισμού. Αυτό οι 20 συμφωνίε ε, πρέπει να είναι ιδιαίτερα φιλόδοξε από βερλινδική σκοπιά και θα πρέπει να δείξουν ότι θα πετύχουν του στόχου πολιτική πιο φτηνά ή πιο γρήγορα από ό,τι υποχρεωτικέ ρυθμίσει. Αν ε, μπορούν να το κάνουν αυτό, τότε δυνάμει τη οδηγία, ε, δηλώνοντα η προτιμόμενη επιλογή. Η οδηγία θέτει κάποιε προποθέσει που πρέπει να γίνουν σεβαστέ από οποιαδήποτε ακουσία συμφωνία και επικεντρώνεται ιδίως στη διαφάνεια και στο επίπεδο φιλοδοξίας της συμφωνίας. Ένα τμήμα του λόγου για τι χρήσει ε, των ακουσίων συμφωνιών είναι ότι είναι πιο ευέλικτε ε, και όχι τόσο βαριέ όπω οι κανονισμοί, αλλά παρόλα αυτά και η διαδικασία τη ε, σύναψή του και τη κύρωσή του είναι αρκετά πολύπλοκη. Πρέπει να γίνει ευρία διαβουλευσή με του stakeholders, μελέτη αντικτύπου, στενή παρακολούθηση με τα κράτη-μέλη και όλοι πρέπει να διασφαλίσουν ότι η εθελοντική συμφωνία έχει προσθεμένη αξία. Σε πραγματικό χρόνο, αν ε, δεν πετύχει αυτή η συμφωνία, η Κομισιόν ε, διατηρεί το δικαίωμα πρωτοβουλίας της να έρθει με έναν ε, δεσμευτικό κανονισμό και η πρώτη, και αυτή η συμφωνία αυτή για τους σύνθετους αποκατοικητές θα είναι η πρώτη που θα υιοθετηθεί στα πλαίσια τη οδηγία του οικολογικού συνδυασμού, σύνθετοι οικοδημητέ, κανεί δεν έχει ακούσει τον όρο αυτό, αλλά όλοι το έχουν. Πρόκειται για του δέκτε, για την ψηφιακή τηλεόραση πληρωμή. Περίπου 60 εκατομμύρια απολύθηκαν πέρσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύουμε ότι χωρί τη δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε η συνολική κατανάλωση ηλεκτρική ενέργεια ε, από αυτού θα αυξηθεί διπλασιαστεί. Ξέρετε, ε, ουσιαστικά μπορεί να καταναλώσουν τόσο όσο ένα μικρό ψυγείο και ε, συνεχώς ε, ε, νέες απαιτήσει ε, για ε, την κατανάλωση. Τώρα, εμείς αποφασίσαμε για τρεις λόγους να έχουμε τέτοια ακουσία συμφωνία. Καταρχήν, η ενεργειακή κατανάλωση των σύνθετων αποκοδικητών δεν εξαρτάται μόνο από το σχεδιασμό τους, ε, που είναι αυτό που μπορούμε να επιτύχουμε με τον κανονισμό, αλλά και από το πώς τις γυρίζονται οι εταιρείε ε, και η δυναμική τους μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ε, την εμπλοκή ε, του παρόχου των υπηρεσιών. Αυτό λοιπόν θέλουμε να το πετύχουμε την εθελοντική συμφωνία. Επίση, οι λειτουργίε του εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα και έτσι χρειάζεται μία πιο ευέλικτη προσέγγιση ε, για το να θέτουμε τι απαιτήσει και οι πιο πολύπλοκε τεχνικέ προδιαγραφέ των αποκωδικοποιητών ε, ουσιαστικά ε, γίνεται από εμπειρογνωμένου και έτσι είναι πιο εύκολη η παρακολούθηση. Ε, μαζί με την ε, ήδη την ακούσια συμφωνία, το Κοινοβούλιο κατέληξε ότι η πρόταση της βιομηχανίας αυτή την ακούσια συμφωνία παρέχει το ίδιο επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας που θα είχαμε με τον κανονισμό και Έχουμε και ταχύτερη εκτέλεση. Έτσι λοιπόν πληρεί τι απαιτήσει του παραρτήματο 8 τη οδηγία που έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια και την εμπλοκή τη κοινωνία των πολιτών και επίση προσφέρει καλύτερο δυναμικό βελτίωση μεσοπρόθεσμα μέχρι το 2015 από ό,τι μπορούμε να πετύχουμε το κανονισμό. Και αυτή η δυναμική θα μπορούσε να πληρωθεί αν ε, σιγουρέψουμε ότι όλα αυτά θα τεθούν σε εφαρμογή από τη βιομηχανία και από τα κράτη-μέλη. Ξέρω ότι πολύ συχνά εκφράζονται ανησυχίε για τι συμφωνίας, όμως σε αυτή την περίπτωση δεν δίνουμε λευκή επιταγή στη βιομηχανία. Η πρώτη περίοδος για την υποβολή εκθέσεων ε, λήγει αυτό το μήνα, κατόπιν θα υπάρχουν οι προθεσμία δύο μηνών ε, για να ε, κατατεθούν στοιχεία από τους ανεξάρτητους επιθεωρητές και στο φόρουμ διαβούλευσης, όπου συμμετέχουν και τα κράτη-μέλη αλλά και οι διάφοροι συμμετέχοντες θα συζητηθούν όλα αυτά το φθινόπωρο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς το λόγο για το σημείο αυτό, τους συναδέλφους. Όχι. Οπότε μπορούμε να κηρύξουμε το πέρα της συνεδρίασης με θερμές ευχές για καλές διακοπές. Οι επόμενε μας συνεδριάσεις θα γίνουν στις 8 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, 3 με 6,5 και 12 Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο από 7 και 4 μέχρι 9 παρατέταρτο. Σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι και είστε επανειδήν το Σεπτέμβριο.